Καλημέρα σας. Άρχεται η συνεδρίαση. Ε, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έχουμε την ε, δήλωση της Επιτροπής σε σχέση με την εγκριθής απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο.